On va commencer les travaux. On dit toujours que les absents ont toujours tort, les retardataires aussi. Donc, euh, nous sommes au point 10 de... Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με την Joan Carling, που δραστηριοποιείται στην στην, στον αγώνα της για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Ε, τρία, τρεις ακτιβίστες ανθρωπίνων δικαιωμάτων σκοτώνουν τη βδομάδα σε όλο τον κόσμο, δολοφονούνται. Ε, κυρίως ε, υπερασπίζονται τα δικαιώματα, τα θεωρητικά δικαιώματα, ιδιαίτερα στον κλάδο της, τον τη της δασοκομείας, της γεωργίας και τη εξορρυκτική βιομηχανία κυρίως. Οι αυτόχθονοι λαοί, οι ηθαγενεί λαοί βρίσκονται στο κέντρο του προγράμματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, μέχρι το 2030. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της βιοποικιλότητας βρίσκεται στα εδάφη τους. Ήδη έχουμε μια έκθεση για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Υιοθετήσαμε αυτό το ψήφισμα τον Ιούλιο του 2018. Ε, καλωσορίζω λοιπόν την Τζοάν Κάρλινγκ αγωνίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ε, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αυτοκτόνων λαών και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Ε, θα ήθελα να τη εκφράσω την υποστήριξή μου όπως και σε όλους τους, ε, σε όλο το λαό στην, ε, στις Φιλιππίνες ο οποίος σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ευάλωτος.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 Yeah, perhaps it's your hat. Yeah. Thank you. Okay. Yes, uh, good morning to uh, to everyone, and I, I sincerely appreciate this. Uh... Καλή σας μέρα. Χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση. Είναι η πρώτη μου παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που μας έχετε δώσει και ιδιαίτερα ε, στον τον τυφώνα που έπληξε την ε, χώρα μας, που είναι και αυτό ένα από τα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Να σας ε, παρουσιάσω την κατάσταση των Ιθαγενών λαών γενικά στον κόσμο και μετά θα σας πω ποια είναι τα βασικά προβλήματα που έχουμε εμείς στις Φιλιππίνες και θα δούμε μετά μαζί στη συζήτηση πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ηθαγενών λαών με την αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων μας και την συμπερίληψή μας στην, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Οι αυτόχθονες λαοί αντιπροσωπεύουν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, κάτι παραπάνω δηλαδή από 400 λαοί το 15% αυτών είναι πάρα πολύ φτωχοί. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αναλφαβητισμού σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα το 80% της ε, βιοπικιλότητας του κόσμου βρίσκεται σε περιοχές αυτοχθονών λαών. Περιοχές που αντιπροσωπεύουν το 60% της γης, ενώ το μόνο το 10% αυτό να έχει αναγνωριστεί από τον νόμο. Γι' αυτό το λόγο προκαλούνται και οι συγκρούσεις ε, για την γη των αυτοχθών λαών, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε κατοχυρώσει τις γης μας. Τι είναι οι αυτόχθονοι λαοί, λαοί σε σχέση με τις μειονότητες ας καταλάβουμε ότι ε, στην ιστορικά, να δούμε ιστορικά τη δημιουργία των αυτοχθόνων λαών. Αν δείτε την παγκόσμια ιστορία, την απεικιοποίηση και τη δημιουργία κρατών, υπάρχουν, υπήρχαν κοινότητες ε, επιτόπου πριν την, τον απικισμό. Κοινότητες οι οποίες είχαν θεσμούς, κουλτούρα και ταυτότητες. Οπότε όταν έγινε η απικιοποίηση, ο απικισμός και δημιουργήθηκαν απικιοκρατικά κράτη, αυτές οι κοινότητες σε ένα μεγάλο βαθμό αποφάσισαν να διατηρήσουν τις, ε, την ταυτότητά τους, την κουλτούρα τους, τους δεσμούς τους, τα όργανά τους, την οργάνωσή τους και την άμεση και στενή σχέση με τη γη τους και με τους πόρους που βρίσκονταν εκεί, τους φυσικούς πόρους. Αυτή η διάκριση, αυτή η διαφορά, αυτή η επιμονή μας κάνει αυτό που είμαστε σήμερα. Θέλουμε να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τη γη μας και τις ε, ταυτότητές μας, ε, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τον τρόπο ζωής μας σε σχέση με το, την κουλτούρα την οποία ε, δημιουργήσαν τα κράτη. Οπότε, βασικά μας χαρακτηριστικά είναι αυτή η σχέση μας με τη γη. Ε, δεύτερον, ότι το ταυτοποιούμαστε ως αυτόχθονες λαοί. Τι θα πει αυτό, ταυτοποιούμενοι. Ε, νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα, σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Και αυτή είναι η διαφορά από τις μειονότητες. Οι μειονότητες μπορεί να έχουν κάποια θρησκεία, κάποια συγκεκριμένη κοινωνική πρακτική, αλλά δεν έχουν ε, εθιμικό δίκαιο και συστήματα που τους ενώνουν. Δεν έχουν αυτή την αλληλοεξάρτηση με τη γη τους και με τους φυσικούς πόρους. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αυτοκτών λαών και μειονότητων. Εγώ έχω εργαστεί στην Ασία για 8 χρόνια και η, ε, στην Νοτιοανατολική Ασία οι αυτόχθονες λαοί μπορούν να ονομάζονται εθνικές μειονότητες οι εθνοτικές μειονότητες ε, και αλλά υπάρχουν και άλλες λέξεις σε άλλα μέρη της Ασίας. Παρόλα αυτά όλοι αυτοί είναι αυτόχθονες λαοί γιατί αυτό έτσι ονομάζουν τον εαυτό τους. Τώρα ένα κράτος μπορεί να τους ονομάσει εθνοτική μειονότητα. Στην πραγματικότητα όμως οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται αυτόχθονες ή ηθαγενείς λαοί και έτσι θα πρέπει να τους θεωρούμε. Έχουν με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα τα οποία αναφέρει η δήλωση του, η διακήρυξη του ΟΗΕ ε, του 2007 για τα δικαιώματα των αυτοχθών λαών. Επιστρέφοντας στην ιστορική αφήγηση. Ο Οργανισμός Ομένων Εθνών ε, κατέδειξε και προέβαλε αυτή τη διαφορά και έδωσε ε, στους αυτόχθονες λαούς ε, διάφορα δικαιώματα μόνο με αυτόν τον τρόπο, με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορούμε να επιβιώσουμε ως αυτόχθονες λαοί. παρά την υιοθέτηση της διακήρυξης του ΟΗΕ, παρά την ύπαρξη μηχανισμών του ΟΗΕ για τα δικαιώματά μας, για παράδειγμα έχουμε το Μηχανισμό Εμπειρογνωμών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθών Λαών και το Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίση έχουμε το μόνιμο φόρουμ για θέματα ε, αυτοχθών λαών στη Νέα Υόρκη και έχουμε και τον ειδικό εισηγητή για τα δικαιώματα των αυτοχθών λαών. Όλοι αυτοί οι θεσμοί, όλα αυτά τα όργανα εξετάζουν το πώς τα κράτη προστατεύουν και αναγνωρίζουν τα δικαιώματά μας. Η δυσάρεστη όμως πραγματικότητα είναι ότι ε, τα δικαιώματα, η κατάσταση των δικαιωμάτων χειροτερεύει, επιδεινώνεται. Βλέπουμε όλο και περισσότερες παραβιάσεις αυτών. Και κυρίως γιατί ε, της ύπαρξης ε, αυταρχικών κρατών. Στις Φιλιππίνες η νομοθεσία για τα δικαιώματα των αυτοκτών λαών είναι αυστηρή, αλλά όλο και περισσότερο ε, παραβιάζουν τα δικαιώματά μας επειδή οι γέες μας πουλιώνται σε Κινέζους και σε άλλους επιχειρηματίες. Και μάλιστα μερικές φορές αυτό γίνεται στο όνομα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, μας αφαιρούνται Μα αφαιρείται η γη μα στο όνομα της βίωσιμη ανάπτυξη ή ε, με την δικαιολογία ότι αυτό θα αποτελέσει λύση στην κλιματική αλλαγή. Αυτό το φαινόμενο ε, είναι επιδεινούμενο σε πολλές χώρες. Μερικές ε, φορές οι υγιές αφαιρούνται από τους αυτόνου λαούς για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις με την με την αιτιολόγηση ότι θα προστατευτούν, θα προστεθούν δηλαδή σε φυσικά πάρκα ε, τα οποία δημιουργούνται ε, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής που υποτίθεται θα πρέπει να οδηγήσει σε, σε ε, προστασία και συντήρηση μας αφαιρούνται οι μας γιατί θεωρείται ότι εμείς δεν μπορούμε να τις προστατεύσουμε. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά οπωσδήποτε στην Ασία. Η συνεχιζόμενη έλλειψη αναγνώρισης των δικαιωμάτων των αυτοχθών λαών νομικά οδηγεί και σε διώξεις εναντίον μας, γιατί υπάρχουν νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν παραδοσιακά μας επαγγέλματα όπως το κυνήγι, ε, η αμυψή σπορά, ε, η, η συλλογή ξύλων, καρπών, μελιού κλπ. Εκατοντάδες ε, δικοί μας άνθρωποι είναι στις φυλακές για αυτούς τους λόγους. Το δεύτερο είναι ότι μας αφαιρείται η γη μας και όταν εμείς ε, διαμαρτυρόμαστε, κατηγορούμαστε για τρομοκρατία ή λένε ότι ε, εμποδίζουμε την ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση η δικαιοσύνη στρέφεται όλο και περισσότερο εναντίον μας. Όταν προστατεύουμε, όταν προασπιζόμαστε τη γη μας, μας απευθύνουν κατηγορίες ε, για καταστροφή διοκτησίας, ε, μας κατηγορούν ότι εμποδίζουμε την ανάπτυξη, όπως είπα μόλις πριν. Στο Βιετνάμ για παράδειγμα, ορισμένες από τις εθνοτικές μειονότητες καταγγέλλονται ε, ότι δρούν ενάντια στο εθνικό συμφέρον. <laughs> δεν κατανοούν ότι οι άνθρωποι δεν βγαίνουν στον δρόμο έτσι τυχαία, μόνο και μόνο επειδή θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Βγαίνουν στον δρόμο και διαμαρτύρονται ή ε, διαδηλώνουν όταν η ζωή τους και το βιός τους κινδυνεύει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα θέμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όταν ποινικοποιείται μια πράξη, μια διαδικασία, ε, τι, μπορεί να, τι μπορεί να κάνει αυτό αυτόν λαοί. Το δίκαιο αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτέ οι επιχειρήσει χρησιμοποιούν τι άδειέ του, τα συμβόλαιά του, τι συμβάσει που έχουν και λένε ότι έχουν δικαίωμα να λειτουργήσουν. Ναι, <laughs> λειτουργούν όμω και δραστηριοποιούνται σε γη αυτοκτών λαών και το δικαίωμα των αυτοκτών λαών στη γη του δεν αναγνωρίζεται. Αυτό ονομάζουν οι χώρε αυτέ κράτο δικαίου. Δεν μπορεί να είναι κράτο δικαίου όταν δεν ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. γιατί αυτό το κράτος δικαίου προσπίζεται τα συμφέροντα μόνο ορισμένων των επιχειρήσεων και όχι των αυτοχθόνων λαών. Τα συλλογικά μας δικαιώματα παραβιάζονται. Οπότε η ποινικοποίηση των αυτοχθόνων λαών αυξάνεται, επιδεινώνεται. Και μάλιστα με τα αυταρχικά καθεστώτα και με τους νόμους για την εθνική ασφάλεια οι οποίοι ε, υιοθετούνται όλο και περισσότερο οι αυτόχθονες λαοί και οι ακτιβιστές τους κατηγορούνται ότι είναι τρομοκράτες και αυτό οδηγεί σε δολοφονίες αλλά και σε συλλήψεις, ε, βασανισμούς κλπ. Υπάρχει και το θέμα των γυναικών. στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, ακόμα και στη Βόρεια Αμερική, το trafficking, το εμπόριο γυναικών από αυτόχθονες λαούς αυξάνεται. Στην Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά πάνω από 10.000 αυτόχθονες γυναίκες είναι εξαφανισμένες και οι περισσότερες είναι θύματα του trafficking. Και στην Ασία το βλέπουμε αυτό, το εμπόριο ανθρώπων συμβαίνει στο Ινμιανμάρ, στο Βιετνάμ ακόμα και στο Βιετνάμ, στην Ταϊλάνδη ε, στέλνουν τις γυναίκες ως παραδουλεύτρες ή βοηθού βοηθούς στην Κίνα. Και κανείς δεν το καταλαβαίνει, κανείς δεν το καταγράφει. Πολλέ γυναίκες αυτοκτόνων λαών δεν έχουν καν υπηκότητα. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν εξαφανιστούν, κανείς δεν τις ψάχνει διότι δεν υπάρχουν για κάποια χώρα. Επίσης δεν λαμβάνουν εκπαίδευση, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, οπότε γίνονται αμέσως πιο ευάλωτες στην εκμετάλλευση και στην παρενόχληση, στην κατα... σε καταχρήσει κλπ. Στο Καμερούν, για παράδειγμα, ή στο Μπουρούντι, πάνω από το 50% των αυτοχθόνων δεν έχουν νομική αναγνώριση, δεν έχουν υπηκότητα δηλαδή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί ανισότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Έχω χρόνο. Ωραία. Πρώτον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έχει κάνει σε σχέση με τους αυτόχθονες λαούς. Έχετε εκδώσει αρκετά ψηφίσματα και πραγματικά σας ευγνωμονούμε ε, για όλα αυτά τα ψηφίσματα που προσπίζονται τη γη μας και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Για παράδειγμα, το ψήφισμα ε, του Κοινοβουλίου, το περσινό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και αυτό για την ε, διαφανή διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο. Και στο ζήτημα της ε, μείωσης της ε, το οποίο είναι ένα πρόβλημα σημαντικό και επίκαιρο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαστε το τέταρτο χρόνο και ο ΙΕ, ε, ο λέει ότι έχουμε μείνει ήδη πίσω σε όλες τις χώρες. Στην Ασία δε η κατάσταση χειροτερεύει. Για παράδειγμα, στο περιβάλλον η αποψήλωση των δασών, η μείωση της βιοποικιλότητας, η μόλυνση, όλα αυτά χειροτερεύουν, όλοι οι δείκτες αυτοί χειροτερεύουν. Σε ό,τι διαφορά το κεφάλαιο 16 για την ειρήνη και τα δημοκρατικά, τους δημοκρατικούς θεσμούς, ακόμα και οι δημοκρατικοί θεσμοί υφίστανται επιθέσεις, όλο και μεγαλύτερη ποινικοποίηση, όλο και περισσότερες παραβιάσεις, όλο και περισσότερες συγκρούσεις για τους για τους αυτόχθονους λαούς δε υπάρχει και το πρόβλημα της έλψης πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Αυτό το ζήτημα ε, είναι κεντρικό σε όλες τις ε, συστάσεις των οργάνων του ΟΕΕ. Έλλειψη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάσεις ε, των δικαιωμάτων στους πόρους και τη γη τους ε, και παραβιάσεις το δικαίωμα πληροφόρησης και γνώμης. Όλα αυτά τα αναφέρουν στις αιτήσεις εκθέσεις τους τα όργανα του ΟΗΕ και αν μπορούσαν να διορθωθούν αυτά θα είχαμε πρόοδο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αν δεν εντάξουμε πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στο, στη ρητορική μας για την ανάπτυξη, ποτέ δεν θα καταφέρουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να ε, επιτύχουμε την ανάπτυξη χωρίς να αποκλείσουμε κανένα, χωρίς να αφήσουμε κανένα πίσω. Ακόμα και στη συμμετοχή, αν δεν συμμετέχουν οι πολίτες στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, πώς είναι δυνατόν να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των κατόχων των δικαιωμάτων, των δικαιούχων. Θα πρέπει δηλαδή η προσέγγιση μας να είναι από κάτω προς τα πάνω για την εφαρμογή των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όχι από πάνω προς τα κάτω. Και για τους αυτόχθονες λαούς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε αφανείς. Παρόλη την σημαντική μας παρουσία σε πολλές χώρες και παρόλη τη συνεισφορά μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, εμείς διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τους πόρους. Το, το δικό μας, ο δικός μας τρόπος ζωής έχει το χαμηλότερο ε, ίχνος διοξιδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου. Ακόμα και στην, στην ε, ατζέντα που έχουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην άλλη ε, για την κλιματική αλλαγή, ακόμα και εκεί, στις δύο αυτές ατζέντε, ε, στα δύο αυτά θεματολόγια, αγνοούμαστε και η συμμετοχή μας είναι ελάχιστη. Δεν μας δεν μπορούμε λοιπόν να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μετάβαση που χρειάζεται να γίνει ε, για να προστατευτεί ο πλανήτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, Ιζαμπέλ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας που ήταν τόσο γαλήνια. Είπατε πράγματα τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν. Είναι δύσκολα πράγματα, αλλά τα είπατε με τρόπο που μπορούσαμε να σας παρακολουθήσουμε πλήρως. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Ήταν σαφή αυτά που είπατε. Θα ήθελα να ρωτήσω απλώς τι εσείς περιμένετε από μας. Γιατί ξεκάθαρα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο Εσεί τι νομίζετε ότι μπορούμε εμεί να κάνουμε για εσά. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για του Σοσιαλδημοκράτε. Ιζαμπέλα. Τίμους. 5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υπεύθυνο για το 80% της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί μας ε, δείχνει το πραγματικό βάρος ε, των αυτοκτών λαών στην προστασία ε, του πλανήτη και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, στην ε, προστασία της βιοποικιλότητας. Ένας Γουαρανί από τη Βραζιλία λέει ότι <laughs> υπάρχει πολύ γη για λίγους Ινδιάνους της Αμερικής, αλλά είναι λίγοι Ινδιάνοι της Αμερικής για να προστατεύσουν όλο τον πλανήτη. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ανεξαρτήτως αυτού βλέπουμε ότι λαμβάνει η χώρα με πραγματική τεράστια επίθεση εναντίον των αυτοχθών σε όλο τον κόσμο. Ε, εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη τους πολλές φορές, ε, διώκονται, δολοφονούνται. Η κυρία Κάρλινγκ μίλησε για διάφορα ε, μέσα στο διεθνές νομικό στερέωμα, στη διεθνή ανομητάξη και πιο συγκεκριμένα στα όργανα του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Τι, τι είναι αυτό που δεν πάει καλά στην προστασία αυτών των αυτοκτονών παρόλο ότι έχουμε τόσα όργανα, ε, τόσους μηχανισμούς. Είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, είναι ε, η απονομή της δικαιοσύνης, είναι η πρόθεση μέτρων προστασίας, σαφών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας. Τι είναι αυτό που δεν δουλεύει, που έχουμε αποτύχει, γιατί ο αριθμός των δολοφονιών, των ανθρωποκτονιών, ε, οι διώξεις εναντίον ε, μελών των αυτοκτών λαών ε, αυξάνονται ε, με τρόπο που μας τρομάζει. Τι δεν λειτουργεί λοιπόν σε θεσμικό επίπεδο, όχι μόνο στις χώρες, αλλά κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Μια και εμείς είμαστε τμήμα αυτού του διεθνούς επίπεδου. Μιλήσατε για τους, τα διάφορους θερμούς και τους διάφορους μηχανισμούς του ΟΗΕ. Αν ακόμα και έτσι δεν μπορούμε να καταφέρουμε να περιορίσουμε ε, το φαινόμενο και αντιθέτως βλέπουμε όξυνση των προβλημάτων, κάτι δεν πάει καλά. το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, κυρία Κάρλινγκ. Όταν ε, μιλάμε για τους αυτόχθονες ε, πληθυσμούς, ε, σκεφτόμαστε πληθυσμούς που βρίσκονται εκτός Ευρώπης κυρίως. Υπάρχουν όμως αυτόχθονες πληθυσμοί και εδώ στην Ευρώπη. Και είχα τη χαρά να πάω στην Νορβηγία και τη Ρωσία πέρσι και συνάντησα πληθυσμούς Σάμι. Αναρωτιόμουν λοιπόν εάν ε, μπορούμε να δούμε εδώ κάποιο μοντέλο, το οποίο σίγουρα δεν είναι τέλειο και μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά οι Σάμοι μετά από μακροχρόνια πάλι κατόρθωσαν να έχουν τουλάχιστον τη δική τους βουλή, στην Νορβηγία τουλάχιστον. Βεβαίω, η Νορβηγία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι κάτι παρόμοιο έχει γίνει και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Ε, με τους Σάμι και άλλους ε, ε, αυτόχθονες. Μπορείτε λοιπόν να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα όπου έχει γίνει πρόοδος. Πώς θα θέλατε λοιπόν ίσως ε, σε διεθνές επίπεδο να είναι οι σχέσεις με τις κυβερνήσεις και πώς μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του παραδοσιακού τρόπου ζωής αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονα στους αυτόχθονες να προοδεύσουν, να βγουν από την φτώχεια τους. Μπετίνα. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε γιατί μας ε, αναφέρατε με αρκετά παραδείγματα κάποια πράγματα για τα οποία είμαι ήδη πεπισμένη δηλαδή ότι με... μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αυτόφωνες λαούς όσον αφορά την διαχείριση των πόρων που ζουν με έναν τρόπο που είναι πολύ αηφόρος και δεν καταστρέφει τον κόσμο θεωρώ ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι όλες οι δηλώσεις του ΟΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα ψηφίσματα γενικώ είναι αποτελεσματικά μόνο αν είναι νομικά δεσμευτικά στο εθνικό δίκαιο. Και εκεί αποτυγχάνουμε συχνά. Και αυτός είναι ένας λόγος ε, για τον οποίο ε, στις περισσότερες περιπτώσεις αγνοούνται τα δικαιώματα των αυτοχρόνων. Και συχνά αυτό σχετίζεται με πόρους που βρίσκονται στις περιοχές όπου ζουν. Παραδείγματος χάρη ε, υπάρχει η σχετική συμφωνία του ILO η παριθμόν 169 για την προστασία των αυτοχρόνων λαών, η οποία έχει κυρωθεί από ελάχιστα κράτη. Λοιπόν, πάρα πολύ συχνά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λένε καλά λόγια και κατηγορούν τους άλλους, αλλά όταν μιλάμε στην αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης ή της προστασίας από την αρπαγή γης, μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τίποτα και αποτυγχάνουν. Λοιπόν, Υπάρχει ένα κομμάτι, κάτι κάνουμε ευτυχώς, αλλά πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα έτσι ώστε κατά μήκο των παγκοσμίων εφοδιαστικών αλυσίδων να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπάρχει μια πιστοποίηση ότι αυτά γίνονται σεβαστά. Αλλά κατά την άποψή σας, ποια είναι ε, η σημαντικότερη πρωτοβουλία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ε, κατάστασή σας. Κάποιο άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Εγώ θα είχα να κάνω μια ερώτηση. Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν κάποιες βέλτιστες ε, πρακτικές ε, όσον αφορά την συνύπαρξη ανάμεσα στους αυτόχθονες πληθυσμούς και τους ε, άλλους πληθυσμούς, της πλειοψηφίας όπως λέμε, όσον αφορά την χρήση των πόρων, του εδάφους, της γης. Υπάρχουν τέτοια καλά παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν στο μέλλον για τις μελλοντικέ μας εργασίες εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, αλλά και για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από τις παραβιάσεις, γιατί συνεχίζονται και τι πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως, το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά. Ο λόγος για τις παραβιάσεις είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους των κρατών για την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων κυρίω όσον αφορά την προστασία των πόρων, διότι βεβαίω εμπλέκονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα όσον αφορά τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ και ποιε από αυτέ απομένουν ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι περισσότερε υπάρχουν σε εδάφη αυτοχθόνων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρου των κρατών για να προστατευθούν αυτέ οι γέε. Και υπάρχουν χώρες που έχουν νόμους, οι οποίοι όμως παραβιάζονται. Και βεβαίω υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις, οι που είναι εταίροι κυβερνήσεων σε πολλά κράτη. Υπάρχει φαρπαγή γύσα Και πολλές φορές θυσιάζεται η βιοπικιλότητα για το κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν και ο ιδιωτικός τομέας, οι μεγάλες επιχειρήσεις, ε, να αρχίσουν να σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και να προστατεύουν το περιβάλλον. Γιατί χωρίς βιωσιμότητα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει ο πλανήτης. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι σήμερα. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε προστατευτικά μέτρα για την αηφορία, δεν θα τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανισμούς. Όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειάζεται λογοδοσία αποτελεσματικοί μηχανισμοί λογοδοσίας, τόσο για τα κράτη όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Χωρίς αυτή τη λογοδοσία μπορούν ε, να τη γλιτώνουν ε, συνέχεια αυτές οι επιχειρήσεις ε, και τα κράτη, ακόμα και με φόνο. Και βεβαίως υπάρχουν και οι φαρπαγές γης, οι εξώσεις πληθυσμών, οι εκτοπισμοί πληθυσμών. Γι' αυτό ακριβώς τα πράγματα χειροτερεύουν σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για βιωσιμότητα όταν οι ανισότητες αυξάνονται συνεχώς. Όταν ε, κάποιοι ε, μέσα στην κοινωνία εκμεταλλεύονται τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ισχυρότερους μηχανισμούς λογοδοσίας και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Διότι χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς θα συνεχίσουν δυστυχώς ...η παραβιάσεις. Και θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε δράση κατά των απολυταρχικών καθεστώτων, να έχουμε περισσότερο δημοκρατικό περιθώριο, να προστατεύσουμε τους ε, προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν δεν τους υποστηρίξουμε. Εάν δεν τους στηρίξουμε, κανένας δεν θα το κάνει. Αυτή η ατιμορρησία θα συνεχιστεί επάπειρον. Και βεβαίως υπάρχουν ε, παραδείγματα, υπάρχουν ε, ε, καλές περιπτώσεις προστασίας έγκυων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες και υπεράσπισης των υπερμάχων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ψηφίσματα και θα πρέπει όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε τελικά. Διασφαλίζοντας ότι υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ότι υπάρχουν μηχανισμοί στήριξης για τα θύματα της σα και για τις οικογένειές τους. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. είναι ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε και πολλά άλλα διαφορετικά όργανα. Έχετε και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έχετε και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε λοιπόν να δούμε, για παράδειγμα, πώς το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να επιβλέψει ε, τον αντίκτυπο ε, του εμπορίου. Συμπεριλαμβάνοντας και τις μεγάλες εταιρείες. Διότι ναι, γίνονται καταστρατηγήσεις, ξεκάθαρα. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μου. Όπου έχει γίνει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταστρατηγήσεις στο πλαίσιο της σύμβασης που, έχει υπογράψει, που έχουν υπογράψει οι Φιλιππίνες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ ε, σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να δράσουμε προορατικά. Η σύσταση λοιπόν που έχει ήδη ε, διατυπώσει το Ευρωκοινοβούλιο προς τον ειδικό εισηγητή είναι η επίβλεψη για να δούμε πως οι δεσμεύσεις προς τους αυτόχθονες πληθυσμούς πραγματικά εκπληρούνται. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και κάτι άλλο που εμείς θα θέλαμε να προτείνουμε, επίσης προορατικό μέτρο, είναι το Ευρωκοινοβούλιο να εξετάσει έναν μόνιμο διάλογο με τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Να δημιουργηθεί ένας τέτοιος διάλογος για να συζητείτε η πρόοδος αλλά και το πώς οι δραστηριότητες ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο τον κόσμο επηρεάζουν τη ζωή των αυτοχθόνων πληθυσμών. Για παράδειγμα, έχουμε την IFAD, το Διεθνές Ταμείο για την Γεωργική Ανάπτυξη. Είναι ένα μόνιμο φόρουμ αυτόχθονων πληθυσμών ε, που συναντάται, σε, ε, ε, συναντάται κάθε δύο χρόνια Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ε, πρακτική σε διεθνές επίπεδο. Διότι έτσι μπορούμε να έρθουμε σε άμεση ε, επαφή με τους ηθήνοντες. δεν θα πρέπει να διαχωρίζουμε την ανάπτυξη από τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών. Δεν θα πρέπει να απομονώνουμε αυτά τα δύο θέματα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί τρόποι να δράσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί επίσης να, μπορούν επίσης να βοηθήσουν για μεγαλύτερη συμμόρφωση όσον αφορά το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πώς όλα αυτά μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένα πώς ε, μπορούν να στηρίξουν περισσότερο τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το Indigenous Navigator που είναι μια πρωτοβουλία για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και έχει σχέση με τους, ε, βιώσιμους, με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Θα ήταν ενδιαφέρον για το Ευρωκοινοβούλιο, νομίζω, να μάθει περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία. Ε, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε 11 χώρες, εκ των οποίων 6 έχουν αναγνωρίσει δια νόμου την έγκαια ιδιοκτησία, τα δικαιώματα. Όμως, παράλληλα, γίνεται ακόμα χειρότερη η φαρπαγή Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε όταν μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται επί τόπου, ε, ποιες είναι οι ζημίες, ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές ε, και την χρήση των πόρων ε, και όσον αφορά το δίκαιο. Μπορεί ίσως να εκπλαγείτε αν μάθετε αυτό που συμβαίνει στην Χιλή, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ προοδευτική ενεργειακή πολιτική όσον αφορά τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Έχουν ε, στην ενεργειακή τους πολιτική και πρωτοβουλίες για ανανεώσιμε ενέργειες. Και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια διαρκής πάλι με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και ότι ο μόνος τρόπος είναι ο διάλογος και να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές. Είναι μια ενεργής ε, συμμετοχή λοιπόν των αυτόχθονων πληθυσμών στην χάραξη της ενεργειακής πολιτικής. Σιγά σιγά λοιπόν υποχωρεί η αντιπαράθεση και τώρα υπάρχει μεγαλύτερη θέληση συνεργασίας αυτοκτόνων πληθυσμών κυβέρνησης για να εφαρμοστεί η ενεργειακή πολιτική. Διότι υπάρχει ανάγκη αυτοί που χαράσουν την ενεργειακή πολιτική να στηρίζουν παράλληλα και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. η ενεργή άμεση συμμετοχή των αυτοχθόνων πληθυσμών στην χάραξη της πολιτικής. Διότι τελικά και τα δικαιώματα και οι φιλοδοξίες λαμβάνονται υπόψη. Και όσον αφορά τους Σάμι, έχετε δίκιο. Υπάρχει Βουλή των Σάμι και στη Φιλανδία και την Σουηδία και συνεργάζονται όλες αυτές οι βουλές μεταξύ τους και υπάρχει και το Συμβούλιο Σάμι που είναι ένα άλλο δίκτυο που συνδέει τους πληθυσμούς Σάμι. Η Βουλή των Σάμι έχει να κάνει περισσότερο με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, αλλά δεν έχει μεγάλη εξουσία όσον αφορά τη γη και τους πόρους. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορούν να θέσουν υποσυζήτηση. στην Φιλανδία υπήρξε μια εξέλιξη όσον αφορά την παραδοσιακή αλληλεία και τους Σάμι. υπήρξαν αποφάσεις σχετικά με την αλληλεία και τον περιορισμό της που αντέβαινε προς τα δικαιώματα των Σάμι. Τουλάχιστον όμως με τη Βουλή τους, οι Σάμι έχουν μία διεπαφή, έναν μηχανισμό για δημιουργία διαλόγου με το κράτος. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί για δημιουργία διαλόγου. Και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργία τέτοιων μηχανισμών, ούτω ώστε οι αυτόχθονε πληθυσμοί από τη μια, το κράτο από την άλλη, να μπορούν ανοιχτά να δημιουργήσουν ένα διάλογο, να συζητήσουν τι υποχρεώσει ε, του κράτου έναντι των αυτοχθόνων. Διότι δεν μπορεί ξαφνικά οι αυτόχθονε πληθυσμοί να εκδιώκονται από τη γη του. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο πλαίσιο πάλι μιας συμμετοχικής δημοκρατίας. Και νομίζω ότι εδώ το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί πραγματικά να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τέτοιους μηχανισμούς, να δημιουργηθεί ένας τέτοιος διάλογος. Και εδώ βεβαίως μπορούν, μπορούν και τα Ηνωμένα Έθνη να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να τις κάλυψα όλες. Ναι, νομίζω ανέφερα ήδη τις ελλείψεις, τη λύπη στην, για την εφαρμογή της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων νομικών μέσων που έχουμε. Ε, ένα πλαίσιο ρυθμιστικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις και δημοκρατική συμμετοχή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Γιατί χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών. δεν μπορούμε να κάνουμε τις κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη τους σοβαρά τις δεσμεύσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω να σας απάντησα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. I'm actually here on behalf of my... Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τους συναδέλφους ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης. Ε, καλώς ήρθατε κυρία Κάρλινγκ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε και τα σημειώσαμε. Είναι πολύ επίκαιρα δεδομένου ότι χτες ξεκίνησε και η 25η Σύνοδος των Μερών στην Ευρώπη και βεβαίως για εμάς ε, τους Ευρωπαίους ε, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που είναι παγκοσμίο αλλά επηρεάζει πλέον πολλούς ανθρώπους στην καθημερινή ζωή τους και αυτόχθονες βεβαίως πλήττονται περισσότερο από τους άλλους Τώρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πω σύντομα το τι κάνουμε. Το γεγονός ότι έχουμε προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων ε, των αυτοχθόνων είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εκπληρωθούν και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και αναφέρομαι και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 2017 για τους αυτόχθονες λαούς όπου η απειλή που υφίστανται ειδικά σχέση με τη φύση και το περιβάλλον είναι κορυφαία προτεραιότητα. Επίση ο δεσμό που έχουν οι άνθρωποι με τη φύση, με το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιβίωσή σα Τώρα, μέσω τη αναπτυξιακή συνεργασία κάνουμε διάφορα πράγματα, δεν μπορώ να αναφέρθω σε όλα. Να πω ότι έχουμε ισχυρού μηχανισμού προστασία για υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε λάβει 30.000 επίγουσε κλήσει και Μία στις τέσσερις από αυτές ε, προέρχεται από υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της γης ε, και μία στις δέκα από υπερασπιστές ε, δικαιωμάτων των αυτοχθόνων. Λοιπόν, φροντίζουμε να ενδυναμωθούν αυτές οι κοινότητες, να ακούγεται η φωνή τους, υπάρχει η σχετική γραμματεία, υπάρχει βεβαίως και ο ο δικό χάρτης αυτός ε, που αφορά 11 χώρες μόνο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα σημαντικό θέμα οπωσδήποτε είναι οι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ζητήσαμε από την ε, κοινωνία των πολιτών να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών για να συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις για να δούμε πώς μπορεί να περιοριστεί ο κίνδυνος ακριβώς από τον αρνητικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω πως έχουμε το 21ο φόρουμ των ΜΚΟ σήμερα και αύριο με θέμα φτιάχνοντας ένα μέλλον για το περιβάλλον για να δούμε πώς θα μπορέσουν οι δράσεις μας ε, να έχουν μεγαλύτερη συνοχή και αντίκτυπο με ε, βεβαίως ε, ιδιαίτερη έμφαση στους αυτόχθονες, τις γυναίκες και τους νέους και θα μιλήσει και εκεί η κυρία Κάρλινγκ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε κυρία Κάρλινγκ και βεβαίως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με σας, με τους αυτόχθονες και βεβαίως η σχέση βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο θέλουμε να έχουμε κατά νου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 11. Ανταλλαγή απόψεων με τον Ομάρ Σακύρ, διευθυντή της Human Rights Watch για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Όπως γνωρίζετε, ο Ομαρ Σακύρ απελάθη πριν από λίγες μέρες από το Ισραήλ. Ήταν εκτελεστικός διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής μάλλον της Human Rights Watch. Δήλωσε ότι το Ισραήλ γινόταν έτσι πρώτη δημοκρατία που απέλασε ένα μέρος της Human Rights Watch. Ο Μαρσακύρ εργάστηκε ε, πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, η κατάσταση στην περιοχή Ισραήλ και Παλαιστίνη σήμερα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι περιοριστικοί νόμοι και ε, η κοινωνία των πολιτών συρρυκνώνεται. Είχαμε την ευκαιρία να το καταγγείλουμε αυτό στην Επιτροπή, μάλιστα αλλά και στην Ολομέλεια κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο. Συνεχίζοντας λοιπόν τις εργασίες μας θεωρήσαμε ότι ήταν χρήσιμο να ακούσουμε σήμερα τον Περιφερειακό Διευθυντή μιας από τις πιο σημαντικές οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Human Rights Watch. Στις 18 του περασμένου Νοεμβρίου, ο Μάικ ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε ότι δεν είναι αντίθετο, όπως είπε προς το Διεθνές Δίκαιο, δεν είναι ε, παράνομη η Ισραηλινή επικισμή. Καλά θα κάνει να ξαναδεί το Διεθνές Δίκαιο. Και η Human Rights Watch κατήγγειλε ότι οι Ισραηλινές αρχές τα μέσα Νοεμβρίου 2018 κατέστρεψαν 390 ε, σπίτια Παλαιστινίων και εκτόπισαν με τη βία 407 πρόσωπα. Πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε εδώ την ε, ε, Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα ε, δικαιώματα του παιδιού. Σήμερα όμως η κατάσταση για τα παιδιά στην Γάζα, αυτά που γεννήθηκαν το 2009, θα έχουν γνωρίσει τρεις πολέμους και στρατιωτική κλιμάκωση και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα και παιδιά που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές σήμερα. Ο Μαρσακίρ τώρα Περιφερειακός Διευθυντής της Human Rights Watch από τον Οκτώβριο του 2016 είναι μαζί μας σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική και στο Ισραήλ δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού. Έχει ξεσπάσει έντονη βία στην Γάζα. Και υπάρχει λοιπόν μια σύραξη χαμηλής έντοσης όπως λέμε, η οποία όμως απειλεί συνεχώς να ξεσπάσει. Κύριε κύριοι έχετε το λόγο. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ο Μάρ Σακύρ λέγομαι. Είμαι διευθυντή για Ισραήλ και Παλαιστίνη στην Human Rights Watch. Πριν από 8 μέρε ε, το Ισραηλινό κράτο με απέλασε επειδή υπερασπιζόμουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά από προσπάθεια 2,5 ετών για να φημώσει την οργάνωσή μας ε, και το κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 όταν η κυβέρνηση του Ισραήλ ε, αρνήθηκε στην οργάνωσή μας, ε, μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, την άδεια να προσλάβει ξένους υπηκόους στο Ισραήλ όταν βεβαίως αυτό γύρισε μπούμεραγκ μετέβαλαν την απόφασή τους και τελικά μας έδωσαν άδεια και μου έδωσαν και εμένα βίζα για να εργαστώ στο Ισραήλ. Την επομένη έφτασα τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησαν νομικές διαδικασίες κατά της οργάνωσης ενώ η αρχική κατηγορία ήταν ότι η Human Rights Watch έκανε προπαγάνδα και όχι, δεν ασχολούνταν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα άλλαξαν το επιχείρημά τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ, το Ισραήλ έφερε έναν φάκελο των μυστικών υπηρεσιών κατά μιας οργάνωσης των δικαιωμάτων και ως εκ τούτου το Μάιο του 2018 διατάθηκε η απέλασή μου και την Δευτέρα μας πέρασε πριν από 8 μέρες αφού εξαντλήθηκε κάθε νομικό μέσο και αφού το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ενέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης ε, και τον νόμο ε, στον οποίο βασιζόταν, αναγκάστηκα να φύγω από το Ισραήλ. Και είναι η πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που βρισκόμαστε στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα που διώχνουν ε, ένα μέλος του προσωπικού μας. Δηλαδή το Ισραήλ πλέον συντάσσεται με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Βενεζουέλα και το Ιράν που έχουν μπλοκάρει την οργάνωσή μας και την πρόσβαση του προσωπικού μας. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να σας πω σήμερα είναι το ότι αυτό το οποίο συνέβη σε εμένα και στην οργάνωσή μας δεν είναι μοναδικό. Έρχεται το μέσο μιας συνεχούς επίθεσης ε, κατά οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λειτουργούν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν μπορέσει να μπουν στο Ισραήλ περιλαμβανομένων ε, βουλευτών από την Ευρώπη και της ειδική ηγήτρια ε, του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα της Παλαιστίνης. Επιπλέον, οι Ισραηλινοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, έχουν υποστεί επίθεση, μεταξύ των οποίων και ο εκτελεστικό διευθυντή ε, τη ε, επιφανέστερη τέτοια οργάνωση, Χαγκάλα, ο οποίο είχε έρθει στο. οποίος κατηγορήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως συνεργάτης του κατακτητή και προδότης. Οι δε Παλαιστίνοι έχουν την χειρότερη μοίρα. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν και αντιμετωπίζουν και ποινικέ κατηγορίες και συλλήψεις τους τελευταίους μήνες μόνο. Ναι, ένας Παλαιστίνιος υπάλληλος της Διεθνούς Αμνηστίας ε, δεν μπορούσε να φύγει από την Δυτική Οχθή για άγνωστους λόγους ασφαλείας. Ε, κάποιος επίσης εργαζόμενος για την Μπέτσελεμ, Ισραηλινή Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, κρατήθηκε τους τελευταίους μήνες ε, η Αντλαμίρ οργάνωση κρατουμένων Παλαιστινιακή υπέστη επίθεση στα γραφεία της από τον στρατό. Η απέλασή μου δε είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Το γεγονός ότι το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ επικύρωσε με την απόφασή του την επίθεση της κυβέρνησης Νετανιάχου στα υπεραστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλεί να συρρυκνώσει ακόμη περισσότερο τον χώρο που έχουν οι υπεραστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ισραηλίνοι και Παλαιστινοί. Η δικαιολογία της κυβέρνησης ήταν ότι ζήτησα μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Η Human Rights Watch ποτέ δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ε, θέση, δεν λαμβάνουμε θέση για μποϊκοτάζ οποιασδήποτε χώρα ή εταιρεία. Αυτό το οποίο κάνουμε και ακούσατε κάποια πράγματα από την κυρία είναι ότι καταγράφουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους πάντες, μεταξύ των οποίων και τις εταιρείε. Και ζητάμε από τις εταιρείε, όπως ζητάμε και από τα κράτη, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ δηλαδή απλά βασικά πράγματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα οποία κάνουμε σε 100 χώρες ανά τον κόσμο. Αυτά τα οποία κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα στην ε, Μέση Ανατολή και στην ε, Βόρεια Αφρική. Και για αυτά τα βασικά πράγματα ε, διέταξαν την απέλασή μου. Η Ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις κατηγορίες για στήριξη στο κίνημα μποϊκοτάζ του Ισραήλ για να επιτίθεται στους υπερασιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2011 επέτρεψε έναν νόμο που επιτρέπει τις μηνύσεις κατά υποστηρικτών του μποϊκοτάζ του Ισραήλ και το 2017 τροποποίησε την νομοθεσία για να απαγορεύεται η είσοδο στη χώρα σε αυτούς και σήμερα στο τέλος του 2019 απελάβνει έναν υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οργάνωση του οποίου δεν έχει θέση για τα μποϊκοτάζ. Ε, για θέματα δηλαδή ε, ειρηνικής έκφρασης. Πού, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους. Σήμερα η κατηγορία αφορά το μποϊκοτάζ του Ισραήλ, αλλά το σκεπτικό του δικαστηρίου βασίστηκε στο ότι το να επιτίθεται κανείς στην νομιμότητα των οικισμών που είναι νομίζω θέμα συνένεσης ε, σε όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται σήμερα σε αυτήν την αίθουσα είναι το ίδιο με το να επιτίθεται κανείς στην νομιμότητα του ίδιου του Ισραήλ και το να ζητάμε από άτομα να μην είναι συνένοχα σε αυτήν την παρανομία είναι λόγος απέλασης. Ε, η ίδια λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να μην ε, επιτρέπεται η είσοδος σε ευρωβουλευτές παραδείγματο χάρη που στηρίζουν ε, την απόφαση τη σχετική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να απαγορεύσουν την είσοδο σε όσους ζητάνε από το ποινικό δικαστήριο να ξεκινήσει μια επίσημη έρευνα για τα εγκλήματα που γίνονται στην Παλαιστίνη ή για τα άτομα τα οποία επιμένουν δικαίως ότι η δυτική όχθη είναι κατεχόμενη και όχι αμφισβητούμενη ή ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι και κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο. Εάν η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι οι δραστηριότητες μας ε, είναι κάποιο είδους απειλή προς ε, το Ισραήλ τι μπορεί να τους αποτρέψει από το να επιτεθούν περαιτέρω στους άλλους ε, υπεραστές ανθρωπινών δικαιωμάτων, Ισραηλινούς και Παλαιστινίους που κάνουν την ίδια δουλειά. Μεταξύ των πολλών δηλώσεων στήριξης ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μία δήλωση 23 ομάδων της κοινωνίας των πολιτών του Ισραήλ. και από συνασπισμούς παλαιστινιακών ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο από άλλους ότι αυτός ο πρόεδρος τους απειλεί. Η Ισραηλινή κυβέρνηση φτάνει στα όρια της. Ε, έχει απελάσει έναν εκπρόσωπο ε, μιας οργάνωσης από τις μεγαλύτερες ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά την καταδίκη μεγάλου μέρους του κόσμου. Εάν δεν υπάρξουν συνέπειες τι θα τους εμποδίσει σε λίγες εβδομάδες ή μήνες να αρχίσει να συλλαμβάνει ε, μέλη τέτοιων ανθρώπινων δικαιωμάτων ή να τις εμποδίσει να λειτουργούν. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζεται η διεθνή κοινότητα. Η αξιοψία σας διακυβεύεται. Μιλήσατε και σας αγνόησαν και με απέλασαν. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας. Αυτό θα μας πει πάρα πολλά για το τι θα κάνει μετά η Ισραηλινή κυβέρνηση. Σας ζητάω σήμερα να αναλάβετε δράση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να ζητήσετε από την Ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει την απόφασή της και να μου επιτρέψει να ξαναμπώ στη χώρα. Το Ισραήλ δεν είναι η πρώτη χώρα που διώχνει έρευνητές της ε, Human Rights Watch μπορεί να θέλει μία μέρα να γίνει σαν το Ουσβεκιστάν ή το Κονγκό ή την Αιθιοπία που μετά μας επέτρεψαν να ξαναπάμε στις χώρες. Λοιπόν, να είμαι σαφής. Η δουλειά μας θα συνεχιστεί υπό την διεύθυνσή μου. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση στον κόσμο να έχει βέτο στο ποιος θα κάνει τη δουλειά και τι δουλειά θα κάνει. Ε, αυτοί οι οποίοι βλάπτονται περισσότερο από την απέλασή μου είναι οι εταίροι μας, Ισραηλοί και Παλαιστίνοι, που θέλουν να έχουν την ευκαιρία να είναι σε επαφή με τους διεθνεί διεθνείς ε, συναδέλφους και κυρίως βεβαίως τα θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αξίζουν να έχουν πρόσβαση στους μεγαλύτερους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε η δουλειά μας θα συνεχιστεί, αλλά είναι καλύτερα για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη για τον κόσμο η δουλειά μας να γίνεται εκεί επί τόπου. Το δεύτερο αίτημά μου για προς εσάς και ακόμη σημαντικότερο είναι να διαφυλάξετε έναν χώρο για αυτούς που έμειναν πίσω στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και συνεχίζουν να δουλεύουν. Ήταν βεβαίως πλήγμα η απέλασή μου προς την κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά μας ένωσε κιόλα. και μπορώ να σας πω μετά από δυόμιση χρόνια στην Ιερουσαλήμ σε επαφή με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους συναδέλφους ότι πάντα η κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν ενωμένη και ποτέ δεν ήταν πιο ενωμένη όσον αφορά το κατεπήγον της ε, κατάστασης ε, και για την ε, ανάγκη διεθνούς δράσης όσο τώρα. Ελπίζω λοιπόν να προσκαλέσετε τους Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους συναδέλφους μου να έρθουν εδώ να μιλήσουν και να πάτε να τους επισκεφτείτε και να υποστηρίξετε τη δουλειά τους και να τους χρηματοδοτήσετε. Και υπάρχει και μια προσπάθεια και εδώ στην Ευρώπη για να χτυπηθούν αυτές οι οργανώσεις ε, λέγοντας ότι υποστηρίζουν τον μποϊκοτάζ του Ισραήλ για να φημωθεί η ελεύθερη έκφραση και ο ακτιβισμός. Η περίπτωσή μου να σας υπενθυμίζει όχι μόνο τους περιορισμούς της Ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και τα όσα κάνουν οι υποστηρικτές του Ισραήλ ε, και λένε ότι με προκάλημα το μποϊκοτάζ προσπαθούν να φημώσουν ως κάνουν σοβαρή ανθρωπιστική δουλειά. Και τρίτο και σημαντικότερο, αυτό το οποίο ζητάω από εσάς σήμερα, είναι να ξαναδείτε την προσέγγισή σας όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης γενικότερα. Εάν όλες οι συλλογικές προσπάθειες μας ε, και δηλώσεις μας δεν σταματούν το Ισραήλ από το να απελάσει κάποιον ο οποίο καταγράφει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς θα τις σταματήσουμε αυτές. Οι επιθέσεις στου υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο μιας κατοχής 52 ετών που καθορίζεται από συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεσμικές διακρίσεις. Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά το ότι το βήμα αυτό ήταν άνευ προηγουμένου για την δική μας οργάνωση, έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο διεθνές προσωπικό στη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ εδώ και πάνω από μια δεκαετία και οι υπερασίες ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να βγουν και να μπουν από τη Γάζα. Γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι εδώ και μία δεκαετία το Ισραήλ έχει κάνει την Γάζα μια ανοιχτή φυλακή. Έχει φυλακίσει δύο εκατομμύρια ανθρώπου σε μια λωρίδα γης 40 ε, επί 11 χιλιόμετρα. Δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν φύγει ποτέ από αυτή τη λωρίδα γης. Η προσέγγιση μας λοιπόν ως προς το θέμα της Γάζας έχει αποτύχει και βεβαίως ε, αυτό μας αφορά όλους μας. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ εδρεώνει τους ε, παράνομους ε, επικισμούς. Μιλάμε για 650.000 επίκους αυτή τη στιγμή. Όποτε συζητάμε το θέμα αυτό σε τέτοιους φορείς, συχνά μιλάμε για την ειρηνευτική διαδικασία. Κυρίε και κύριοι, δεν υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία η ειρηνευτική διαδικασία ήταν ένα προκάλημα για να εδρεωθεί μια πραγματικότητα ενός κράτους, μιας μόνιμης κατοχής και άνισων δικαιωμάτων. Ένας Παλαιστίνιος 50 ετών σήμερα στη Δυτική Οχθή δεν είχε ποτέ αστικά δικαιώματα, δεν είχε ποτέ το δικαίωμα να μιλήσει ελεύθερα, να οργανώσει διαδηλώσεις, να ανήκει σε μια πολιτική ομάδα. Έχει γνωρίσει μόνο το καθεστώς το οποίο καθιστά την πρόσβασή του σε βασικές υπηρεσίες, ε, την δυνατότητα να κινηθεί ελεύθερα, όλα αυτά τα καθορίζουμε με βάση το ότι είναι Παλαιστίνιος η θέση των ΙΠΑ τα τελευταία 2,5 χρόνια ξεκαθαρίζει ότι το μπαλάκι πλέον είναι στο γήπεδο της Ευρώπης και σε φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε μια ιστορική ευκαιρία να δράσετε. Η ιστορία θα θυμάται στιγμές σαν και αυτήν. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να πάτε πέρα από τα σύνθηματα, να μην μιλάμε για δύο-τρία κράτη, ειρηνευτικέ διαδικασίες και να δείτε την πραγματικότητα επί τόπου. Μια πραγματικότητα όπου οι Παλαιστίνοι είτε εγκλωβισμένοι στην Γάζα, είτε έχουν κολλήσει σε μια κατάσταση μόνιμης κατοχής ε, και θεσμικής ε, διάκρισης, είτε ως ε, Παλαιστίνοι ε, ω Ισραηλινοί πολίτες να υφίστανται ανισότητα ε, ζουν στην Παλαιστίνη. Η κατοχή συνεχίζεται εδώ και 52 χρόνια. Θα συνεχίσουν να έρχονται άνθρωποι σαν και εμένα να σας λένε τα ίδια και στα 100 χρόνια της ε, κατοχής. Θα σας πω λέγοντας το εξής. Η απέλασή μου και η προσπάθεια εκδίωξης της οργάνωσής μας ε, θα πρέπει ακριβώς να σας οδηγήσει να δράσετε στα ζητήματα αυτά. Η λύση δεν είναι κι άλλες δηλώσεις ή προσπάθειες να υπερασπιστείτε τους ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δείτε το θέμα των ε, παρανόμων, επικισμών και της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι. Δεν θα χάσουμε. Δεν θα σταματήσουμε, με συγχωρείτε την ε, δουλειά που κάνουμε. Απλά ελπίζουμε να είστε στο πλευρό μας και η ιστορία σας παρακολουθεί. Ευχαριστώ. Um, θα ήθελες το λόγο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ομιλία σας, για ομιλία ομιλία πρόκειτο. με πολύ ε, ε, έντιμο τρόπο ε, θα ήθελα να πω ότι δεν αισθάνομαι άνετο όταν μιλάμε για το Ισραήλ γιατί θυμάμαι το πώς δημιουργήθηκε αυτή η χώρα. Δεν μπορώ να μη θυμάμαι το ολοκαύτωμα, τον αντισημιτισμό της εποχής εκείνης που εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα και τους πολέμους, τους οποίους θυμάμαι ως παιδί. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν δικαιολογίες για την σημερινή κατάσταση, για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στα κατεχόμενα εδάφη, την ανισότητα ε, των δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά εισαγωγικά. Τώρα, μίλησατε για την ενευτική διαδικασία. τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν οι Παλαιστίνοι. Γιατί πάντοτε βλέπουμε το θέμα από τη μεριά του Ισραήλ. Έχω την εντύπωση πως χρειάζεται και οι δύο πλευρές να συνεισφέρουν, παρόλο ότι μία είναι πιο ισχυρή από την άλλη. Αν δεν εμπλακούν και οι δύο πλευρές, δεν θα είναι βιώσιμη οποιαδήποτε λύση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των Παλαιστινίων στην επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Μετά, ποιο ρόλο παίζει η αίσθηση του Ισραήλ για έλλειψη ασφάλειας. Εμείς μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο εκεί. Σε Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας. Isabel Santos. Ιζαμπέλ Σάντος. Ήταν πολύ σαφή. Τα λόγια σας και μας διευκρίνησαν το τι συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα προκύπτει από κάποιες δηλώσεις και από κάποιες αλλαγή, αλλαγές πλεύσης ε, της Αμερικανικής κυβέρνησης οι οποίες ε, τροφοδοτούν ε, την αδιαλαξία του Ισραήλ. Η απέλαση αυτή δεν θα είχε συμβεί. Όπως και άλλες παραβιάσεις που έχουν λάβει χώρα τελευταία δεν θα είχαν συμβεί αν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν αποτελούσαν προστάτηδα δύναμη του Ισραήλ. Η διατλαντική συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών πλήττεται από την ε, στρατηγική μετατόπιση των ΗΠΑ τελευταία. Και αυτό έχει και άλλες συνέπειες. Ε, οπότε τώρα ποιος μεριμνά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποιος παρακολουθεί την κατάστασή τους Ποιος προασπίζεται τους ακτιβιστές και τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή την περιοχή. Η έξοδος της Human Rights Watch, η απέλασή σας, ε, είναι ε, αποτελεί ε, επίθεση εναντίον ενός παράγοντα ο οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικός, αξιόπιστος ε, στην περιοχή και ειλικρινά δεν ξέρω τι μένει πια όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη χωρίς την Human Rights Watch πού θα καταφεύγουμε για να ενημερωνόμαστε. Είναι προφανές λοιπόν ότι η αυτή η απέλασή σας επηρεάζει όλη την οργάνωση, αλλά η ερώτηση είναι υπάρχει κάποιος τρόπος να αντικατασταθείτε, να συνεχιστεί η εργασία της Human Rights Watch. Ε, για πάρα πολλά χρόνια γίνονται δηλώσεις από όλες πλευρές, εκκλήσεις και για πολλά χρόνια βλέπουμε ότι αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι εκκλήσεις δεν δίνουν αποτέλεσμα. Πρέπει να περάσουμε σε κάτι πιο απτό. Είναι πολύ ανησυχητή η αύξηση της βίας προφανώς. και ταυτόχρονα θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς η Human Rights Watch σκοπεύει να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, αν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, για να συνεχίσει τις εργασίες της εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Η Ειρήνα. Just, just very briefly and I will also... Θα αφήσω και το συναδέλφους να μιλήσουν, να πω κάτι, δύο λόγια μόνο. Ε, στην την Ισαμπέλ, ε, ως Βρετανίδα ε, αλλά και ως Γερμανίδα, έχω δουλέψει και στη Βρετανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, και είμαι πεπισμένη ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά του Ισραήλ συνεισφέρουν στην αύξηση του αντισημιτισμού. Οπότε από αυτή την πλευρά είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ρυθμιστεί το Παλαιστινιακό και να συνεχίσει να εργάζεται Human Rights Watch εκεί. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ υπάρχει περίπτωση να βελτιώσει την κατάσταση υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού στο Ισραήλ με τις οποίες θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε το διάλογο για να τις θεωρήσουμε συνεργάτες μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κύριε Σάκυρ μαζί μας σήμερα. Τον Αύγουστο επισκέφθηκα την περιοχή με ε, εκκλησιαστικές ομάδες από τη Δανία και ε, συναντηθήκαμε ε, και με Παλαιστίνιους και με Ισραηλινούς και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και αντιληφθήκαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Παλαιστίνοι. Για πρώτη φορά είδα το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην συνδρομή στους έχοντες ανάγκη. Τελευταία ε, ε, ακούμε εκθέσεις ότι το, η, ο νόμος του 2016 του Ισραήλ για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις επιτρέπει στο Ισραήλ ε, να κλείσουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δεν εργάζονται σύμφωνα με τις επιθυμίες της κυβέρνησης του Ισραήλ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη συνέπεια στο έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι Ισραηλινές αρχές έχουν κάνει επιδρομές, ε, μη ανώσεις, έχουν συλλάβει πολλούς αγωνιστές και έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε άλλους. Ε, είδαμε ότι οι πολιτικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από άλλες ε, χώρες έχουν την απαγορευτή είσοδο τους στη Γάζα. Όλα αυτά ε, συμβαίνουν, μαζί με ε, στιγματισμό και λασπολογίες ε, ενάντια σε πολλούς αγωνιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την άποψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν τη βάση της δημοκρατίας και θα αγωνιστούμε για να ακούγεται η φωνή τους. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να ε, εντείνει την στήριξή της σε, αυτούς, σε αυτές τις ορανώσεις με χρηματοδότηση ε, μέσω ε, των μηχανισμών που διαθέτουμε. Δυστυχώς κύριε Σάκερ, η δική σας περίπτωση είναι συμβολική, δείχνει τη συρρήκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και είναι από τέλεσμα της εφαρμογής ε, μιας πολιτικής ατζέντας ε, του συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντα του Ισραήλ που υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία. Τι στήριξη μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εσά, κύριε Σάκηρ, ε, στην οργάνωσή σα, αλλά και γενικότερα στου αγωνιστέ για, τα, για τα δικαιώματα των Παλαιστίνων σε όλο τον κόσμο. Ε, εσείς μας ζητήσατε να ζητήσουμε από το Ισραήλ να ε, ε, αναστείλει την απόφαση του για την απέλασή σας. Ε, πέραν αυτού, αν δεν ξαναξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και των επικισμών, αλλά και γενικότερα του Παλαιστινιακού. Yeah, welcome Mr. Shakir and Thank you that you are here, uh, but I will speak in... Ευχαριστώ κύριε Σακύρ και ευχαριστώ που ήρθατε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη πράγματι δείχνει την απίστευτα δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το Ισραήλ. Ε, βεβαίως ε, δεν είναι δημοκρατική συμπεριφορά γιατί δεν συμβιβάζεται με τις αρχές ε, του κράτους δικαίου και ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε τη σημαντική δουλειά που κάνετε και σας ευχαριστώ για αυτό το οποίο κάνετε και θεωρώ ότι όπως ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ακολουθούσε μία λύση δύο κρατών δεν θα το δεχτεί ποτέ το να υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας όπως ε, περιγράψατε και θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους βεβαίως η Ευρώπη έχει μία ιστορική ευθύνη για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εβραϊκού λαού και στην ε, πατρίδα μου στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο εγώ είμαι υπέρ ακριβώς ε, του να θυμόμαστε το τι συνέβη στο Στάιρμαρκ. Ακριβώς όμως ε, για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Όπως είχε πει και ο Γιτζάκ Ραμπίν, πρέπει να προτιμήσουμε την οδό τη ειρήνη, από την οδό του πολέμου, λίγο πριν δολοφονηθεί. Και τώρα μα λέει ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό ο δρόμο. Οπότε έχω κάποιε σύντομε ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα είχα πάει. Προσφάτως στο Ισραήλ συναντήθηκα με εκπροσώπους κυβερνήσεις και εκπροσώπους ΜΚΟ και μου εξήγησαν την ε, κατάσταση και βεβαίω υπήρχε και το θέμα της οικοδόμησης των οικισμών οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. αυτό το οποίο συμβαίνει και δημιουργεί γεγονότα στο θέμα των επικισμών επιτρέπει να υπάρξει μια λύση δύο κρατών ή τα γεγονότα αυτά πλέον έχουν εδρεωθεί τόσο ώστε δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Και δεύτερον, έχουμε τον επιθετικό πόλεμο της Τουρκίας στην ε, Βόρεια Συρία. Αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχει επηρεάσει την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ. Και η αλλαγή πολιτικής του Ντόναλτ Τραμπ τι, πώς έχει επηρεάσει τους ε, λαούς περιοχής, ε, τις ελπίδες και τις προσδοκίες Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Πώς το βλέπουν αυτοί, ε, πώς βλέπουν την πολιτική του Ντόναλτ Τραμπ. Σας ευχαριστώ κύριος Μοχάμετ. Ναι, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κάποιος ο οποίος πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θεωρώ ότι κανένα κράτος ε, δεν θα πρέπει να βαθμολογεί εαυτό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό ισχύει και για τη χώρα μου το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή πρέπει πάντα κάποιο απ' έξω να μας λέει το τι κάνω και νομίζω ότι η απέλασή σας είναι ένα βήμα προς τα πίσω πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα Ε, αναφέρατε επίσης ε, ε, δύο πράγματα. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι η ειρηνευτική διαδικασία, εάν δηλαδή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση ενός κράτους. Από εδώ και μπρος λοιπόν, πώς βλέπετε τα ανθρώπινα δικαιώματα να εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό και οι ανθρώπους σαν και εμάς, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να ζητήσουμε εάν η λύση των δύο κρατών ε, την οποία συζητάμε τα τελευταία 20 χρόνια δεν είναι πια πραγματικότητα. Τι πρέπει να ζητάμε, τι πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπενιάν. Ναι. Μετά και τις προηγούμενες ερωτήσεις θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι Κοιτάξτε, το κόμμα μου είναι σαφώς υπέρ της λύσης ε, των δύο κρατών, αλλά στην πράξη σε ποιο βαθμό είναι ακόμα δυνατόν να υπάρξει κάποια ανταλλαγή γεών ε, και εάν γίνει κάτι τέτοιο ε, θα πρέπει βεβαίως να υπάρξει και μια αποζημίωση. Αυτό το οποίο βλέπουμε με τους οικισμούς είναι αρπαγή γης αντί για κάποια υποχρεωτική αγορά με αποζημίωση. Οπότε τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος ε, ανταλλαγής ε, γεών για να δημιουργηθεί μια λύση των δύο κρατών ε, όταν θα έχουμε και μια κυβέρνηση στο Ισραήλ η οποία θα θέλει κάπως περισσότερο τον συμβιβασμό και εάν δεν συμβεί αυτό αν πηγαίνουμε σε μια κανονική λύση ενός κράτους ε, θα έλεγα αν δούμε το τι συνέβη σε χώρες όπως η Νότια Αφρική θα καταλήξει να είναι ε, ένα κράτος με βάση ε, ο καθένας να έχει μία ψήφο και μάλλον αυτό δεν θα άρεσε στο Ισραήλ θα προτιμούσαν μία λύση δύο κρατών Οπότε ουσιαστικά είναι ε, η ίδια ερώτηση. Απλά ε, προσθέτω ε, κάποια επιπλέον σημεία συζήτησης. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Θα την κάνω στα γαλλικά. Έχουμε υπενθυμίσει το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε ε, και μπορούμε να είμαστε και ακτιβιστές και ευρωβουλευτές ταυτόχρονα. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι για το σεβασμό του δικαίου και τον έλεγχο αυτής αυτού του σεβασμού. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ επιβλέπει. Ο ΟΗΕ έχει αποφανθεί ότι σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο οι οικισμοί, οι οικισμοί είναι παράνομοι στα κατεχόμενα. Ε, αυτή τη στιγμή και το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείες παραβιάζουν αυτή τη διεθνή νομοθεσία. Ποιε είναι οι δικέ μας δυνατότητε να επιστρέψουμε στην εφαρμογή του δικαίου και ποια μέσα διαθέτουμε. Ε, ένα μέσο που διαθέτουμε είναι η Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει ότι το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβονται μερικά πράγματα μεταξύ αυτών τους νόμους και το δίκαιο, του διεθνού, το διεθνές δίκαιο ή τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα, στο θέμα τη σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από τους, οικισμού. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί και αυτά έχουν το, την υποχρέωση να σεβαστούν το δίκαιο, τι συστήνετε εσείς ως Human Rights Watch στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια, να κάνουν προκειμένου να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο σε θέματα σήμανση, για παράδειγμα. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και για τις ερωτήσεις σας, πολύ, καλή, πολύ καλές ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα. Να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις καταρχήν. Για το θέμα των λύσεων στο οποίο αναφερθήκατε πολύ από σας. Τη συζήτηση της λύσης των δύο κρατών και εμείς δεν υποστηρίζουμε κάποια θέση ως Human Rights Watch που δεν είμαστε ουδέτεροι. Όταν όμως γίνεται λόγος για τη λύση των δύο κρατών, ε, μερικές φορές ε, ξεχνάμε ποιο είναι το πρόβλημα. Συνήθως οι λύσεις προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα, όμως το πρόβλημα πολύ συχνά αγνοείται στη συζήτηση για το, το, τη λύση των δύο κρατών. Ε, το πρόβλημα δεν είναι η οικισμοί, ο επικισμός κλπ. Ε, το, τα δύο κράτη έχουν πλέον χάσει την έννοιά τους γιατί ε, η ύπαρξη δύο κρατών δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα. Ε, σήμερα έχουμε ένα κράτος στην πραγματικότητα το οποίο και πάλι δεν είναι λύση. Οπότε γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις. Συμπεριλαμβανομένων και αυτών τις οποίες αναφέρατε. Αλλά καμία δεν βασίζεται στην αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και των δύο, και Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Το, ε, εν μέρη, το πρόβλημα με την ειρηνευτική διαδικασία είναι το εξή ότι ορισμένοι υπονοούν ότι το πρόβλημα είναι η μη διαπραγμάτευση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί μπορεί να διαπραγματεύεσαι ε, παορίστο και παρόλα αυτά να μην βρίσκεις λύση. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να πιεστούν οι δύο μεριές να βρουν μια πολιτική λύση. Και μια οποιαδήποτε ε, ε γενική ρύθμιση του προβλήματος το ότι δύο εκατομμύρια άτομα από τη Ρωσία της Γάζας δεν μπορούν να ταξιδέψουν, δεν μπορούν ε, τέτοιου είδου προβλήματα δεν μπορούμε να περιμένουμε να τα λύσουμε όταν λύσουμε συνολικά το πρόβλημα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, το Ισραήλ σκοτώνει ε, τη λύση των δύο κρατών. γιατί τελικά έχουμε καταλήξει με βάση τις πράξεις του Ισραήλ να έχουμε τρεις δυνατότητες. Ή η απέλαση των Παλαιστινίων, ή ίσα δικαιώματα σε όλους, πράγμα το οποίο το Ισραήλ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει διότι δεν έχει κάποια τέτοια πρόθεση. Και η τρίτη λύση είναι το apartheid που μπορεί ήδη να έχει εγκαθιδρυθεί. Το Ισραήλ προσπαθεί να αποφύγει να κάνει μια επιλογή. Θέλει ε, και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο. Ε, ε, σας λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει κατοχή. Ε, πώς είναι το να μην υπάρχει κατοχή όταν οι Παλαιστίνοι δεν έχουν τα δικαιώματά τους. Είμαστε πολύ μακριά από μια πολιτική λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εξαναγκάσουμε ε, αυτούς που παραβιάζουν τα δικαιώματα των Παλαιστίνων να αναρωτηθούν για αυτά τα θέματα και να δώσουν μια απάντηση. Κάποιοι μου λένε τι ζητάς. Ζητώ μια συντονισμένη διεθνή δράση που θα ξεπερνάει τις δηλώσεις. Να σας δώσω παραδείγματα. Συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων που μπορούν να αναλυθούν. Πρώτον, όλοι μας θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τον το για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην ε, δημοσίευση ενός καταλόγου επιχειρήσεων που λειτουργούν σε παράνομους οικισμούς. Αυτό δεν έχει σχέση με το κίνημα μποϊκοτάζ ε, από επενδύσεις και κυρώσεις, το BDS. Ε, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στην Μιανμάρ ήδη. Το έχει κάνει η Κομισιόν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, λειτουργούν εκεί. Δεύτερον, θα πρέπει να στηρίξουμε τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο οποίος πολύ σύντομα θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει μια επίσημη ανάκριση για τα ε, εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στην Παλαιστίνη. Ε, αν αποφασίσει κάτι τέτοιο η εισαγγελέα, θα δεχθεί επιθέσει και θα πρέπει να τον στηρίξουμε. Τρίτον, το, Ευρωπαϊκό, το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικέ εβδομάδε μα υπενθύμησε ότι είναι υποχρέωση των κρατών μελών να μην επιτρέπουν στο Ισραήλ ε, να να μεταμφιέζουν ε, προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί στους παράνομους οικισμούς σαν να είναι προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί στο Ισραήλ. Αυτό είναι παράνομο. Θα πρέπει επίσης να λογοδοτήσουν για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων και θα πρέπει κάποιος να δώσει λόγο τι συμβαίνει στη Γάζα και κάθε κράτος θα πρέπει να ε, ε, αρνηθεί ε, να αναγνωρίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα του Ισραήλ στους οικισμούς και στα κατεχόμενα. Αυτό είναι υποχρέωση των κρατών μελών. Νομική τους υποχρέωση. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένες πράξεις που μπορούν να αναλυθούν. Εμείς που βρισκόμαστε εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μακριά από το να αρχίσουμε διάλογο για τη λίστα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δικαιωμάτων καταρχήν. Μετά, ο ρόλος των Παλαιστινίων ας πω ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επίσης ε, παραβαίνει συστηματικά δικαιώματα, ε, για παράδειγμα αφαίρεται συλλήψεις και βασανισμούς, ε, η Χαμάς ε, ξαπολύει πυράβλους και ρουκέτες προς το Ισραήλ και όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους. Αυτό το έχω δει και ε, την τελευταία φορά που είχα επισκεφτεί την Ευρώπη ε, ε, είχα μιλήσει σε, για την ανάγκη να μην χρηματοδοτούνται αυτές οι βίες ενέργειες. Θα πρέπει όμως, θα πρέπει και στις δύο πλευρές να είμαστε βέβαιοι ότι δεν, επιβε... συνεισφέρουμε στην παραβιάση δικαιωμάτων. Η πολιτική όμως για την Γάζα δεν είναι καν πολιτική ασφάλειας του Ισραήλ. Ενώ ε, υπάρχει μια απόλυτη ε, απαγόρευση εισόδου-εξόδου ε, από την Γάζα με εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Ε, κάποιοι ας πούμε μπόρεσαν να βγουν για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά δεν κατάφεραν να ξαναβγούν όταν χρειάστηκε για να πάνε σε ένα συνέδριο. Συνεπώς, η λογική πίσω από τον αποκλεισμό της Γάζας δεν είναι, ε, συλλογική, ε, δεν είναι λογική ασφάλειας. Ε, κάθε κράτος έχει δικαίωμα να πάρει μέτρα για την ασφάλειά του. αν πούν ότι εμείς απαγορεύουμε την είσοδο την έξοδο συγκεκριμένων ανθρώπων για λόγους ασφαλείας, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί έχουν κάνει το τάδε, το τάδε κλπ, θα το δεχόμασταν, ε, θα μπορούσαμε να το προσβάλλουμε. Ε, αλλά ε, η πολιτική του Ισραήλ ε, αφορά όλους τους Παλαιστινίους της Γάζας. Είναι μια πολιτική η οποία είναι πολιτική πλήρους αποκλεισμού. Για την τρομοκρατία να πω ότι η Human Rights Watch θα συνεχίσει να δουλεύει. Οπότε ε, ελπίζω να συνεχίσετε να κοιτάτε το site μας. Ε, έχουμε ε, μια ολόκληρη ομάδα από Παλαιστινίους και Ισραηλινούς που εργάζονται επί τόπου με δικές μου οδηγίες. Εγώ και στην Αίγυπτο και στη Συρία και στο Μπαχρέιν έχω δει ότι έχω, έχω υποστεί απαγορεύσεις εισόδου, οπότε ξέρουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, στην, στο Ισραήλ στις δύο τελευταίες εκλογές ε, συζητήθηκε το θέμα ορισμένων πτυχών αντιδημοκρατικών τάσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, ε, δεν έγινε λόγος για την στρατιωτική κατοχή για τα τελευταία 52 χρόνια. Ε, ακόμα και το Λικούντ, ε, το, η αντιπολίτευση του Νεστανιάχου ήταν υπέρ της απελασής μου. οι επιθέσεις εναντίον ομάδων υπεράσπιση δικαιωμάτων ε, οφείλονται ε, και στην κάλυψη των ΗΠΑ. Ε, οι Ισραηλινοί ε, σας λένε κατά βάση ότι ό,τι δηλώσει και να κάνετε εμείς τις γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια και δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Οπότε είναι ελεύθεροι να επιτεθούν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εγώ ε, μετά για τις συστάσεις σας είπα ε, ποιες είναι οι, οι συστάσεις μου. Σας είπα να συναντηθείτε με τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου. Είναι άνθρωποι πραγματικά ε, ε, αποτελούν ελπίδα για το μέλλον και έμπνευση για αγώνα. Οπότε όταν πάτε να τους συναντήσετε για την ε, ασυμβατότητα της απόφασης αυτής με τη δημοκρατία, με τις δημοκρατικές αρχές. Να πω, να προσθέσω ότι οι δημοκρατίες δεν απελάβουν ε, αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και δεν χρησιμοποιούν πολιτικά κριτήρια για να επιτρέψουν κάποιον να μπει ή να μην μπει ή να απαγορεύσουν κάποιον να μπει σε μια χώρα. Οι δημοκρατίες Ε, είναι ε, η εξουσία του λαού και όχι ενός ανθρώπου επί των υπολείπων. Τώρα, για την πολιτική των πολιτιών Υπάρχει κάτι θετικό εκεί, διότι η πολιτική των πολιτών ε, συσπήρωσε τον κόσμο για θέματα ε, προσφύγων, Παλαιστίνων προσφύγων, για θέματα ε, επιθέσεων εναντίον ε, του, των των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε ε, η συμμαχία αυτή μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου δείχνει το δρόμο για τον υπόλοιπο κόσμο. Και πρέπει όμως να κάνουμε κάτι έτσι. Τέλος, για, και πάλι για το θέμα του ενός των δύο κρατών. Ο, η Human Rights Watch δεν έχει άποψη για αυτό το θέμα, εντάξει. Είμαστε αγνωστικιστές, αλλά όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε οποιαδήποτε πολιτική λύση. Αν οι Ισραηλινοί αποδώσουν ε, πολιτικά δικαιώματα στους Ισραηλινούς από τη μια μεριά του δρόμου, θα πρέπει να δώσουν τα ίδια δικαιώματα και στους Παλαιστίνου στην άλλη μεριά του δρόμου. Ε, αν ε, οι Ισραηλινοί έχουν 24 ώρες τη μέρα ηλεκτρικό, έτσι πρέπει να έχουν και οι Παλαιστίνοι. Εδώ και 50 χρόνια ελέγχει το Ισραήλ και κυβερνά σε αυτά τα μέρη, οπότε θα έπρεπε να έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η πρόεδρο, θέλω να δώσω το λόγο στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Αμάσα Κύρ για την παρέμβασή του. Ξέρετε βεβαίως ότι έχουμε γνώση εδώ και πολλά χρόνια των δραστηριοτήτων της Human Rights Watch σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδίως στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Και πολλές επαφές μας με τον κύριο Σακύρο, όπως είπε και ο ίδιος, τον τελευταίο καιρό είχε να κάνει με παραβιάσεις ε, εκ μέρους και των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Νομίζω ότι συναντηθήκαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, θα ξαναδοθούμε και το απόγευμα και επίσης ε, με εκπροσώπους των κρατών μελών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι βεβαίως κυρία Σακύρα, έλαβα υπόψη αυτά που είπατε για τις ε, δηλώσεις και τις πολιτικές δηλώσεις, αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αντιπροσωπεία μας ε, στο Τελαβίβα παρακολούθησε από κοντά την υπόθεση του κυρίου Σακύρ, ε, συμμετείχαμε και στην, ε, παρακολουθήσαμε και τη δίκη, συναντηθήκαμε με τους δικηγόρους του κυρίου Σακύρ και με τις πρεσβείες των 28 κρατών μελών στο Ισραήλ και ε, είχαμε σημαντική δράση, κάναμε δηλώσεις και από τις Βρυξέλλες τον Μάιο, τον περασμένο Μάιο και άλλη μια πριν από λίγες εβδομάδες. Βεβαίως, όπως υπόθηκε, είναι ε, μέρος της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η στήριξη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπως πολλοί είπαν εδώ σήμερα, και όπως φάνηκε ξεκάθαρα και από τις σχετικές δηλώσεις, Στηρίζουμε το ε, δικαίωμα ελεύθερη έκφρασης, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και του συναθρίζεστε και το δικαίωμα των ε, ε, οργανώσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων να δραστηριοποιούνται παντού και στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Το κάναμε στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση του εις του κυρίου Σακύρ και για να μπορέσει έτσι η Human Rights Watch να συνεχίσει το έργο της. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις ε, οργανώσεις των πολιτών ε, και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη παρά τις πολυάριθμες επιθέσεις που δέχονται. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε, Ομάρ. Ελπίζουμε ότι θα λάβεις και πάλι την άδεια να επιστρέψεις και να συνεχίσεις το έργο σου στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Γιατί σε χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη Human Rights Watch εκεί, όπως ήδη είπαμε. Και ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσεις τη δουλειά σου. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για το έργο σου. Περνάμε στο τελευταίο σημείο του σημερινού μας, της σημερινής μας πρωινή συνεδρίασης, την αποστολή στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην Ιζαμπέλ Νομίζω η Ιζαμπέλ Σάντος βγήκε. Θα δώσω το λόγο στην Ειρήνα για να κάνει ένα μικρό απολογισμό. Δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα σε όλη την αποστολή. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Ειρήνα κατευθείαν. Θα σας κάνει την παρουσίαση. Ειρήνα, αν προτιμάς, αν θέλεις μπορούμε λίγο να περιμένουμε ένα λεπτάκι για να φύγουν αυτοί που θέλουν να φύγουν. Λοιπόν, η Ειρήνα, έχεις ε, τον λόγο. Ευχαριστώ, λέει η Ειρήνα. Πόση ώρα μπορώ να μιλήσω. Εσύ λοιπόν θα κάνεις αυτή την περιληπτική παρουσίαση, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω μια σύντομη αναφορά για την κοινή μας αποστολή αφετ Ντρόι σεντε στα Ηνωμένα Έθνη και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Συμμετείχαν ε, εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Θα επικεντρωθώ κυρίως στις συναντήσεις που είχαμε εμείς από τη δική μας Επιτροπή. Θα σας κάνω λοιπόν μια σύντομη περίληψη ε, του τι αποκομίσαμε από αυτές τις ε, συναντήσεις που είχαμε. Και βεβαίως αν θέλετε μπορώ να σας δώσω επιπλέον ε, πληροφορίες, ε, περαιτέρω λεπτομέρειες ε, σε όποιον ενδιαφέρεται. Για μένα τα κυριότερα σημεία είναι πρώτον στα Ηνωμένα Έθνη όπου πήγαμε καταρχάς ότι όσον αφορά την πολυμερή προσέγγιση υπάρχει μια κρίση σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει ένα κενό από την αποχώρηση των ΙΠΑ από τα πολυμερή φόρα, κυρίως όσον αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε πολιταρχικά καθεστώτα όπως τη Ρωσία και την Κίνα να καταλάβουν αυτό το κενό, να μπουν στη μέση και αυτό το έκαναν ε, επανειλημμένος με κάποια σχετική επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται σήμερα ο πιο σημαντικός πυλώνας πολυπλευρικότητας σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο υπάρχει αίσθηση ότι συρρυκνώνεται ο χώρος για τις ΜΚΟ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει έντονη πόλωση, μερικές φορές ε, φτάνει σε αδιέξοδο, παρόλο που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν ε, ε, δρούν αποτελεσματικά. Δεν ξέρουμε πόσα θα συμμετέχουν στο μέλλον, ίσως να είναι μόνο μία ε, χώρα που θα συμμετέχει στο μέλλον ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Η Δύση γενικά με τον Τραμπ στη ΣΥΠΑ έχει χάσει έδαφος και επιρροή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. και όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να δείξουμε, να είμαστε πιο θαραλέοι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Σας έκανα μια περίληψη από την επίσκεψή μας στα Ηνωμένα Έθνη. Επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο της ε, συνέλευσης ε, καταρχάς ε, και συζητήσαμε για τις προτεραιότητες, για την κλιματική αλλαγή και για μια ενδεχόμενη συνεργασία, μια εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά με εκπροσώπους του Αντώνιο Γκουτέρος, του Γενικού Γραμματέα, ήταν μια πολύ ε, καλή συνάντηση. Μάλιστα συναντήσαμε και τον ίδιο τον κύριο Γκουτέρες. Ε, μιλήσαμε για συμπεριληπτικότητα, για πολυπλευρικότητα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας είπε και το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό ότι η καταστρατηγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν σήμερα στην αύξηση της τρομοκρατίας και ότι θα πρέπει στην πάλι κατά της τρομοκρατίας να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως, τρομοκρατία συζητήθηκε ε, επανειλημμένος κατά τη συνάντηση, αλλά θα ήθελα να τονίσω αυτά που μας είπε. Μας είπε ότι η πάλι ε, κατά των εξτρεμισμών συνδέεται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπε ότι τα περιθώρια στενεύουν για την κοινωνία των πολιτών και ότι τα απολυταρχικά καθεστώτα οθούν ε, τον κόσμο ε, σε, στα άκρα και τον εξτρεμισμό. Ε, πολλά άλλα υπόθηκαν, αλλά ήταν τα σημαντικότερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπως είπε και η Ιζαμπέλ Σάντος, μάλλον όπως θα σας πει και η Ιζαμπέλ Σάντος, την αφήνω να συμπληρώσει ότι ενδεχομένως ξέχασα. Αυτά, Μαρία, εκ μέρους μου. Α, επίσης συναντήσαμε και τον αρμόδιο για την ε, Ευρώπη και την Λατινική Αμερική. Επίσης έγιναν κάποιες συζητήσεις και από αυτή την πλευρά, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Και με τους πρέσβεις των Ηνωμένων Εθνών, κύριο Κόλ και κυρία Τσάλι, που μας ε, μίλησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την απόσυρση των Ηνωμένων από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μας είπαν ότι αυτό ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας θέτει ε, επανειλημμένως θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από πλευράς είπα, αυτή η απόσυρση ήταν απαραίτητη και όπως μας είπαν θεωρούν ότι αυτό έχει σχέση και με την ε, Βενεζουέλα. Επίσης αναφέρθηκαν και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και την Σαουδική Αραβία. Συμμετήσαμε επίσης ε, τον Γενικό Γραμματέα κατά της τρομοκρατίας. Δεν έχω κάτι να αναφέρω εδώ. Και τέλος συναντηθήκαμε με την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών Ανιά Καλαμάρ που θα συναντήσουμε σήμερα το απόγευμα. Δεν θα μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες. Ήταν όμως μια πολύ σημαντική συνάντηση. Η κυρία Καλαμάρ μας ενημέρωσε για τις τέσσερις εκθέσεις που συνέταξε για τις γυναίκες, τις μειονότητες, ε, τους ε, μετανάστες και την περίπτωση της δολοφονίας του ε, Τζαμάλ Κασόγγι. Θα μας ενημερώσει περαιτέρω το απόγευμα. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε με τον Ρίτσαρντ Γκάουν, και με την Ινδική Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη και τους πρέσβεις εκεί. Συζητήσαμε πολλά διαφορετικά θέματα, μεταξύ των οποίων η την κατάσταση στο Κασμίρ, η οποία πώς να το πω, τι λόγια να βρω. Ήταν μια εντελώς ανοιχτή, θα έλεγα, συζήτηση. Και δόθηκε πρόσκληση για πρόσβαση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, Βεβαίω όλα αυτά έγιναν τον Οκτώβριο, πολλά πράγματα έχουν γίνει έκτοτε. Στη συνέχεια συναντήσαμε τον Κρίστιαν Μπράουν, πρέσβη. Και που συμμετέχει σε επιτροπή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. για θέματα όπως ρύθμιση, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, το σύμφωνο για τους μετανάστες και πολλά άλλα θέματα. Επίσης, τέθηκε και το θέμα της παραπληροφόρησης. Και μετά είχαμε ένα γεύμα εργασίας με μέλη των Ηνωμένων Εθνών από το Συμβούλιο Ασφαλείας Νομίζω ότι ε, ε, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν περισσότερο την ΑΦΕΤ, τις εξωτερικές υποθέσεις. Είχαμε ένα, όπως είδατε, πολύ βαρύ πρόγραμμα. Μετά συναντηθήκαμε με την κυρία Πάτεν για θέματα βίας ε, στις ένοπλες συγκρούσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και νομίζω ότι υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στη δική της αποστολή και το δικό μας πρόγραμμα, αυτό που έχουμε ε, αποφασίσει για του χρόνου. Η κυρία Πάτεν ανέφερε κυρίως το βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών, ή τουλάχιστον αυτό που απειλεί να θέσει, σε ένα ψήφισμα για τις γυναίκες το 2467 κυρίως για τις γυναίκες της ανώπλες συγκρούσεις. Οι ΙΠΑ δεν είναι ευχαριστημένες με οποιαδήποτε αναφορά στην αναπαραγωγική υγεία και τις αμβλώσεις. Επομένως, προσβλέπουν στην Ευρώπη για να στηρίξει ε, τέτοιου είδους ψηφίσματα. Μίλησαμε επίσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ μπορεί να συνεχίσει κάποιε από αυτέ τι εργασίες και τον συνεχιζόμενο διάλογο που θα έχουμε με την κυρία Πάτεν και νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να επιδιώξουμε να τον συνεχίσουμε. Τέλος, στα Ηνωμένα Έθνη είδαμε τον ε, ε, Μαρκ Λόλοκ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Βεβαίως μιλήσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Πήραμε το τρένο πολύ αργά, στη συνέχεια πήγαμε στη Ουάσιγκτον, όπου είχαμε πολλές διαφορετικές συναντήσεις και οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ε, πραγματικά, ο, μάλλον η επικεφαλής ήταν πραγματικά ε, πάρα πολύ ικανή. Οι συναντήσεις μας έγιναν, διαφορε... έγιναν ξεχωριστά, ξεχωριστά δηλαδή η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ξεχωριστά οι άλλες δύο επιτροπές. Και συναντήσαμε τρία μέλη του Κογκρέσου, γυναίκες, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ η Ιζαμπέλ Βίσλερ, γιατί έχει, είχε μια άλλη συνεδρίαση. Αλλά η Ιζαμπέλ Σάντος και εγώ είδαμε λοιπόν την Γιάννα Πρέσλι, που είναι από τους Δημοκρατικούς, από τη Μασαχουσέτη, και ήταν η πρώτη ε, μαύρη που μίλησε, όπως ε, ίσως ξέρετε, ευθαρσός ε, δέχτηκε επίθεση λεκτική από τον πρόεδρο Τραμπ και εργάζεται κυρίως για την κατάρριξη της θανατικής ποινής και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε ότι ε, αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες πάμε κάπως προς την αντίθετη κατεύθυνση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Όταν όμως μιλήσαμε στην κυρία Πρέσλι υπήρχαν πέντε άτομα τα οποία ε, θα καταδικάζονταν, ε, θα θανατώνονταν σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Συζητήσαμε λοιπόν το θέμα αυτό και μετά της απευθύναμε μία πρόσκληση να έρθει να μας μιλήσει εδώ ε, του χρόνου στο πλαίσιο των συζητήσεών μας για τη θανατική ποινή. Στη συνέχεια είδαμε την κυρία Βερόνικα Εσκομπάρ και αυτή από τους Δημοκρατικούς από το Ελπάσο. συζητήσαμε για την κατάσταση στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού, για την κατάσταση των οικογενειών εκεί. Είχαμε μια ακρόαση εδώ και θα έχουμε επίσης μία το Φεβρουάριο του χρόνου. Νομίζω ότι η συνάντησή μας με την κυρία Σκομπάλ ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Κάποια στιγμή με δάκρυα στα μάτια μας μίλησε για τις οικογένειες αυτές πάνω στα σύνορα και μας είπε ότι χωρίστηκαν 1.500 οικογένειες περισσότερες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί. Προσπαθούμε λοιπόν ε, με την κυρία Εσκομπάρ να συνεργαστούμε για να ε, διευκολύνει την αποστολή μας στη μελλοντική στο Ελπάσο. Τέλος, είδαμε την κυρία Ντίγκελ, επίσης ε, από τους Δημοκρατικούς, που εργάζεται κυρίως για τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους και την ενδοοικογενειακή βία. Ήταν ίσως η πιο πρόθυμη από τη, τα τρία μέλη του Κογκρέσου που συναντήσαμε να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί μας, ίσως σε πιο θεσμικό επίπεδο ε, και να γίνει και μια συνεργασία ανάμεσα στο Κογκρέσο και το Ευρωκοινοβούλιο πάνω σε αυτά τα ε, θέματα. Επίσης, ε, είχαμε μια συνάντηση, ένα γεύμα εργασίας ε, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, συζητήσαμε τη θανατική ποινή, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσει, τους πρόσφυγες και για παράδειγμα, η Freedom House ήταν μία από αυτές τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Συμμετείχε, αλλά και εκπρόσωποι από αμερικανικά πανεπιστήμια. Σας αναφέρω κάποια ονόματα οργανώσεων που συμμετείχαν. Δραστηριοποιούνται όλες αυτές οι οργανώσεις σε αυτούς τους τομείς. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι που σας ενδιαφέρει από όλους αυτούς τους τομείς που ανέφερα και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πείτε το το απόγευμα ήταν νομίζω το αντίθετο από το πρωί εκείνης της μέρας. Πήγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και είχαμε κάποιες κοινέ ε, συνεδριάσεις, συναντήσεις με τον υπεύθυνο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και με τον κύριο Abrams, τον ειδικό εκπρόσωπο για τη Βενεζουέλα συζήτησαμε για πολλά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα. Μετά είδαμε τον Μάικλ Μέρφυ, που είναι υφυπουργό Ασφάλειας και Άμυνας και ενημερωθήκαμε και για θέματα με το Ιράν. Και το πιο σημαντικό ίσως συναντήσαμε τον διευθυντή για τα γυναικεία θέματα που ήταν άντρας και συζητήσαμε για τις διαφορές ανάμεσα στην πολιτική των ΗΠΑ και την ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Και βεβαίως προσεγγίσαμε και το θέμα των αμβλώσεων. Βεβαίως, σε περισσότερα θέματα πρέπει να πούμε ότι ε, συμπίπταν οι απόψεις μας. Επίσης, ο Διευθυντής για τις θρησκευτικές ελευθερίες, επίσης, συναντήθηκε μαζί μας, μιλήσαμε και με αυτόν, ακούσαμε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει μια ετήσια έκθεση πιο συγκεκριμένα για την Θρησκεία. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις μπορώ και εδώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Και τέλος συναντήσαμε τον Ρόμπερτ Ντέστρο που νομίζω ότι θα έρθει εδώ στις 9 Δεκεμβρίου να μας μιλήσει που είναι διευθυντής του Γραφείου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία Μιλήσαμε πιο συγκεκριμένα για τους ε, καταβλισμούς ε, στα σύνορα είπα Μεξικού. Έχουμε κάνει κάποιες ερωτήσεις, δεν έχουμε λάβει ακόμα απαντήσεις. Και ε, επίσης δείξαμε τα θέματα της Κίνας, του Ιράν και του Σουδάν. Ε, τον πιέσαμε επίση για την Σαουδική Αραβία, αλλά δεν νομίζω ότι οι απαντήσει που μα έδωσε ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικέ από αυτού. Και επίσης μιλήσαμε για την αποτελεσματικότητα μια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, ε, η οποία θα ψηφιστεί ίσως, θα περάσει από το Συμβούλιο. Και επίσης μιλήσαμε για την κατάσταση στη Βόρεια Συρία. Τελευταία συνάντηση με δύο ε, εκπροσώπους ε, της ε, αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, πρώην βουλευτές, που προέρχονται από διαφορετικά κόμματα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων, την οποία θα συνεχίσουμε νομίζω και στο μέλλον. Ε, κάτι που συγκράτησα ήταν ο ρόλος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, προστασία κεφαλαίων, καταθέσεων αλλά και στην προστασία μελών της ε, οικογενειών του καθεστώτος της Βενεζουέλας και πιο συγκεκριμένα η Ισπανία ιδιαίτερος ε, αυτό τον, ε, με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν ε, την κυβέρνηση του Μαδούρου ενδεχομένως κάποιες κυρώσεις ή κάτι παρόμοιο με την Global Magnitsky Act των ΗΠΑ θα μπορούσε να εφαρμοστεί και, στις Ηνωμένες, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτά, δεν θα προσθέσω κάτι άλλο. Ίσως η πρόεδρος ή η Ιζαμπέλ Σάντος θα μπορούσαν να προσθέσουν πράγματα. Η Ιζαμπέλ θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Η έκθεσή σου ήταν τόσο λεπτομερής ε, ε, που δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση. Ε, έχουμε πολλά ως συνέχεια αυτής της επίσκεψης στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει για την αρχή του 2020 επίσκεψη η οποία έχει αποφασιστεί από εμά στα σύνορα Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών και σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι μετανάστες, των παιδιών μεταναστών στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικό. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τις ανταλλαγές ε, απόψεων, με τις ανταλλαγές πληροφοριών ε, για τα παιδιά σε ζώνες, ε, εμπόλεμες ζώνες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μια ομάδα εργασίας που κάνει ένα έργο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει και εμάς έτσι ώστε να δούμε το πρόβλημα αυτό στη Συρία το πρόβλημα των παιδιών σε, στην εμπόλυμη περιοχή της Συρίας. Επίσης μίλησες για την ενίσχυση των σχέσεών μας με τα μέλη του Κογκρέσου και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της βίας εναντίον των γυναικών, έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα των γυναικών να γίνουν και να παραμείνουν διεθνή πρότυπα γιατί βλέπουμε ότι το θέμα της ισότητας των γυναικών, της πρόσβασης των γυναικών σε σεξουαλική αναπαραγωγική εκπαίδευση ε, αμφισβητείται, αμφισβητούνται αυτά τα δικαιώματα ε, σε όλο τον κόσμο, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Επίσης, αναφέρθηκε στην άνση με τη Βερόνικα Εσκομπάρ, που επίσης μπορεί να είναι ένα σημείο επαφή για την διοργάνωση της επισκεψής μας τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Το θέμα της ε, θανατικής ποινής επίσης ε, είναι σημαντικό. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, τις δράσεις διαφόρων οργανώσεων της ΗΠΑ για το θέμα της θανατικής ποινής. Ευχαριστώ πολύ και τις δυο σας ε, για όλα αυτά τα στοιχεία. Επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι κοινό με την Επιτροπή ΔΕΒΕ για την κατάσταση των ε, και την προστασία με την κατάσταση των δικαιωμάτων και την προστασία των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Η συνάντηση θα γίνει στο Q... Πού, σε άλλη αίθουσα όμω. PHS. Στο PHS 4Β1. Στο PHS 4Β1. Είναι κοινή συνάντηση, οπότε θα μεταφερθούμε εκεί.